και εγκρίθηκε. Τα πρακτικά της συνεδριάσεως αυτής θα υποβληθούν στο Κοινοβούλιο προς αποδοχή στην επόμενη συνεδρίαση και ε, κατόπιν αυτού θα προωθήσω τα ψηφίσματα τα οποία υπερψηφίστηκαν και κατόπιν ε, μπορώ να